διάταξη είναι η προφορική ερώτηση για την ε, πυρηνική ασφάλεια 25 χρόνια μετά την καταστροφή στο Τσερνομπίλ. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σόνικ που είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό κύριε Σόνικ για να λάβει θέση ο αρμόδιος επίτροπος. Και ευχαριστώ θερμά τον Επίτροπο κ. Τσεφσοβιτς που έχω αποχωρεί. Καλωσορίζω τον Επίτροπο τον Αρμόδιο. Έχετε το λόγο κύριε Σόνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι στην Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θυμάται τα θύματα αυτής της καταστροφής που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία πυρηνική καταστροφή. Η επέτειος αυτή ε, δίνει ένα τραγικό υπόβαθρο μετά το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα. Μάλιστα ε, το δραματικό αυτό ατύχημα έδειξε την ανυμποριά αλλά και την απερισκεψία των, ε, της, των αρχών της Ουκρανίας που προσπάθησαν να κρύψουν από τον κόσμο τις σοβαρές συνέπειες του ατυχήματος του Τσερνομπίλ. Ας θυμηθούμε μερικά στοιχεία η έκρηξη του αντιδραστήρα οδήγησε σε μόλις γύρω στα 100 χιλιόμετρα, 70% ήταν στο, στην Λευκορωσία. Έφτασε μέχρι τη Σκανδιναβία, την Κεντρική Ευρώπη, ραδιενεργά σωματίδια και στην Πολωνία, μέχρι την Ελλάδα και την Ιταλία στην Νότια Ευρώπη. Και μάλιστα ε, εκενώθηκαν ε, γύρω στα 150.000 ε, άτομα από την περιοχή και μάλιστα 220.000 από την ε, Λευκορωσία, την ε, Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία. Μάλιστα η απερίμωση που οδήγησε το πυρηνικό ατύχημα για το περιβάλλον και την ανθρωπίνη υγεία είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Προσπαθούμε ακόμη να δούμε πόσα ήταν τα θύματα, ε, οι νεκροί από το ατύχημα αυτό. Με βάση την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που πέθαναν από καρκίνο μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 9.000 ε, άτομα. Είχαμε 200.000 ε, ε, νεκρούς και από καρκίνο μπορούν να πάθουν, από καρκίνο μπορούν να πάθουν εξαιτία του Τσερνομπίλ, μπορούν να χάσουν τη ζωή του άλλοι 100.000. Ε, μέσα σε δύο ουκρανικές περιφέρειες είχαμε μόλυνση του εδάφους και των τροφίμων. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Ταμείο για το Προστατευτικό Κάλυμα του Τσερνομπίλ και έδωσε μεγάλο αγώνα για να αποτραπούν τα αρνητικά αποτελέσματα του Τσερνομπίλ. Και μάλιστα δώσαμε 100.000 110 ε, εκατομμύρια ευρώ συγγνώμη, ως συμβολή στο ταμείο αυτό του Τσερνομπίλ. Δεν μπορούμε επίσης την 25η επέτειο να ξεχνάμε ότι το θέμα της προσέγγισης της πυρηνικής ασφάλειας είναι ένα διασυνοριακό ζήτημα και παγκόσμιο. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις αρχές της διασυνοριακής υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και να απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κάνουν μακροπρόθεσμες μελέτες ό,τι αφορά τις ε, ε, μακροπρόθεσμες συνέπειες του Τσερνομπίλ. Γιατί θα πρέπει να παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ε, των ανθρώπων τις αρνητικές συνέπειες που είχε το Τσερνομπίλ για την υγεία τους αλλά και για το περιβάλλον. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τέτοια στοιχεία για τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ. Επίσης θα δοθούν νέα κονδύλια προκειμένου να καταπολεμηθούν τα αποτελέσματα του πυρηνικού αυτού ατυχήματος λαμβάνοντα υπόψη τον αριθμό των πυρηνικών εργοστασίων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και το επίπεδο συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πιθανά σενάρια έχουμε σε περίπτωση βλάβη ενό πυρηνικού αντιδραστήρα, ποιε θα είναι οι συνέπειε μια τέτοια βλάβη ε, για του γειτονικού πληθυσμού, υπάρχουν τέτοια σενάρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του συντονισμού. Ε, ε, έχει σχεδιάσει κάποια σενάρια για την εκένωση, σε περίπτωση, εκένωση πληθυσμού σε περίπτωση πυρηνική καταστροφή. Γιατί τέτοια πυρηνικά ατυχήματα δεν έχουν μόνο εθνικέ, αλλά έχουν και παγκόσμιε συνέπειε. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να σκεφτούμε κάποιε αντιδράσει ώστε να ελεγχιστοποιήσουμε του κινδύνου και να αποτρέψουμε τις, ε, τα μεταγενέστερα ατυχήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Ότιγκερ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, στα 25 χρόνια από τότε που συνέβη το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, η Κομισιόν συμμετείχε στις ε, προσπάθειες που αναπτύχθηκαν σε διεθνές επίπεδο για να αμβληνθούν οι συνέπειες του ατυχήματος. Βεβαίω, επειδή πρόκειται για μεγάλο τύχημα, ήταν και απαραίτητο να συνδυαστούν οι δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό συνέβη με ε, κρατημέλη, συνδυασμό ε, δυνάμεων, με τα, την ομάδα G7, με την Ουκρανία. Μεριμνήσαμε λοιπόν έτσι ώστε ο χώρο αυτό ε, να προστατευτεί, να αποκλειστεί, να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέλησε να κινητοποιήσει πόρους έτσι ώστε στο Τσέρνομπιλ να διεκπαιρεωθούν κάποιες εργασίες και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση με δική μας συνεισφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο ε, μεγαλύτερος ε, συνεισφέρον στο Ταμείο για το Τσέρνομπιλ. Ε, τον Απρίλιο είχαμε μια διεθνή διάσκεψη στο Κίεβο για δωρητές και συμβάλαμε με άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ μάλλον συμβάλλουμε άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ και φτάσαμε συνολικά στο ποσό των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, ε, σε διπλωματικό επίπεδο επιτύχαμε 32 χώρες, εκ των οποίων 13 για πρώτη φορά θέλησαν και αυτά να συμβάλλουν ε, με οικονομική χρηματοδότηση σε αυτό το ταμείο. Θα συνεχίσουμε τις ε, δραστηριότητές μας, θα απευθυντούμε και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τους πόρους εκείνους που είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθούν τα προγράμματα μέχρι το 2015. Συνεργαζόμαστε και με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, έτσι ώστε αυτό το έργο της δημιουργίας σαρκοφάγου γύρω από τον χώρο του ατυχήματο να μπορεί να ολοκληρωθεί. Πρόκειται, όπως σας είπα, για, την, για το περίβλημα αυτό. Θα υπάρχει ένα νέο περίβλημα και πρόκειται και για το ότι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να πάψουν να λειτουργούν οι υπόλοιποι αντιδραστήρες. Μέχρι το 2015 προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι εργασίες, το σύνολο του έργου. Κατόπιν στο πλαίσιο του προγράμματος πλαίσιο της Euratom ε, διεξάγονται και άλλες έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνέπειες ε, του ατυχήματος και πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει μια μεγαλεπίβολη πρωτοβουλία, ε, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μελωδία στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πυρηνική ασφάλεια σκεπτόμετα να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα προς όφελος των πολιτών που έχουν πληγεί περισσότερο. Αναφέρομαι στους κατοίκους ε, που ζουν γύρω από το Τσέρνομπιλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ερευνήσουμε περισσότερο τα θέματα της υγείας τους ε, και της διατροφής τους. Ε, εάν λοιπόν υπάρξουν και άλλες ενέργειες που θα αφορούν στην υγεία των πολιτών, αν αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλα μέτρα, η Κομισιόν είναι πρόθυμη να δραστηριοποιηθεί και να αναθέσει στην αρμόδια επιτροπή τον συντονισμό όλων αυτών των ενεργειών. Η αντιμετώπιση λοιπόν της μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι ένα περαιτέρω καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά το ατύχημα συμβάλαμε σε κοινά ερευνητικά προγράμματα ε, τα οποία, ε, στα οποία συμμετέχουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στο να έχουμε καλύτερη διαχείριση πυρηνικών καταστροφών, κυρίως στη Λευκορωσία, στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν στοιχεία σχετικά με την ε, έκκληση ραδιενεργού κεσίου στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το ποινικό ατύχημα. Συγκεντρώσαμε τέτοιου είδους στοιχεία. Το 1998 συγκεντρώσαμε στοιχεία σε συνεργασία με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και την Ρωσία και δημοσιεύσαμε τα στοιχεία αυτά. Αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιο της ε, Euratom ε, στηρίζουμε ένα δίκτυο που αφορά στην ε, ολοκλήρωση, στη διαδικτύωση. Ε, που ε, έχουν σχέση με την ακτινοβολία που μπορεί να πλήξει τους ανθρώπους. Όσον αφορά την πολιτική προστασία, εδώ και εννέα χρόνια ζητάμε να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε ασκήσεις πολιτικής προστασίας, στις οποίες συμμετέχουν και ε, τρίτες, τρίτες χώρες. Αυτά όλα χρηματοδοτούνται από ε, τους δικούς μας τους πόρους για την πολιτική προστασία. Ε, είχαμε το τύχημα, το πλαίσιο το τόρχ, το εκεί στο δεύτερο κυρίως ε, πρόκειται για την περίπτωση μόλυνσης ε, αν εκραγεί ε, βόμβα και ΣΥΜΙΣΕΚ ένα πρόγραμμα όπου πριν από ένα χρόνο έγινε προσωμείωση ραδιενεργούς ενέργειας μετά από σεισμό, έκκλησης ραδιενεργούς ενέργειας. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε με την ευρωπαϊκή βοήθεια να αμπληνθούν δυνατόν οι ζημιές και να αποφευθούν περαιτέρω ζημίες, κυρίως στο χώρο γύρω από το Τσερνομπίλ. Και τώρα εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, πρώτος ο κύριος Ρόιλ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευγνωμονώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας παρουσίασε με τόσο εκτενή τρόπο αυτά τα θέματα και καλό θα ήταν επανειλημμένα να συζητάμε για τέτοια θέματα. Πώς αντέδρασε η Ευρώπη μετά την καταστροφή αυτή άμεσα αλλά και αργότερα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέχρι σήμερα. Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του προβλήματος που είναι ε, μία υπόθεση. Υπάρχει και άλλη υπόθεση που λέγει ότι αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα μέτρα δεν θα είχαν ε, προσλάβει αυτές τις διατάσεις περιορισμού των ζημιών. Επίσης θέλω πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδωσε μόνο έκτακτη επίγουσα βοήθεια αλλά και επιπλέον ως Ευρώπη ασχολήθηκε εντατικά με ε, τα συμπεράσματα και τις επιπτώσεις που θα είχε αυτό ε, στην πολιτική προστασία, στην ανταλλαγή πληροφόρηση, στην έρευνα, στις διάφορες μελέτες. πρέπει να γίνει και μια συζήτηση αν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να έρθουν και νέες μελέτες ή μήπως αυτό που υπάρχει ήδη ως υλικό να ε, το χρησιμοποιήσουμε, να το αξιολογήσουμε, μας αρκεί, είναι αυτό που χρειαζόμαστε, διότι καμιά φορά ε, επειδή υπάρχει πληθώρα μελετών, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο να παραγγέλνουμε και νέες. Ευχαριστώ πολύ και ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρώπη μπορεί να ε, είναι περήφανη με τα όσα έχει κάνει, γιατί δεν μιλάει μόνο, αλλά ε, δρά κιόλα. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, Το λόγο έχει ο κύριος Γιώ Λάινεν. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, κύριε αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ καταρχάς τον συνάδελφο κύριο Σόνικ που ε, κίνησε αυτή τη διαδικασία και την προφορική ερώτηση που οδήγησε στη συζήτηση. Όντω, δεν ε, επιτρέπεται να λησμονούμε την καταστροφή του Τσερλόμπιλ. Ακόμα και 25 χρόνια μετά αυτή την καταστροφή, αυτό τον όλεθρο, είναι μακροχρόνιες οι συνέπειες. Υπάρχει μια μεγάλη περιοχή που ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να επιστρέψει στις αιστείες τους. Ε, υπάρχουν επιπτώσει στην υγεία μακροπρόθεσμες Είχαμε δει ε, και αποβολές 25 ε, χρόνια μετά από την καταστροφή. Οι γυναίκες ε, συνεχίζουν να έχουν προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Και αυτά τα θέματα επίσης της ποινική ασφάλειας δεν είναι θέματα εθνικής κυριαρχίας, αλλά ευρωπαϊκής ευθύνης σε μια ήπειρο που είναι τόσο πύκνο κατοικημένη, κάθε πυρηνικό εργοστάσιο έχει συνέπειες και επιπτώσεις και στο γείτονα. Γι' αυτό, ε, κύριε Τιγκέρ, εσείς φέρετε ιδιαίτερη ευθύνη το θέμα αυτό και με ε, την εμπειρία της Φουκουσίμα ε, χρειάζεται να το χειριστείτε με νέο τρόπο. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με τις δοκιμές ασφαλείας, τα στρέστε των 131 πυρηνικών εργοστασίων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραμείνετε σκληροί στις τάσεις σας. Θέλουμε να έχουμε τα ύψιστα επίπεδα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για τις θεομηνίες να ψάχνουμε ε, και τους άλλους κινδύνους. Ε, να πέφτουν αεροπλάνα, επιθέσεις τρομοκρατικές, επιθέσεις ηλεκτρονικές. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγξουμε κατά πόσο είναι ασφαλείς οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και επίσης ε, να βεβαιωθείτε εσείς να μην είναι μόνο πρόφαση και άλλο αυτό. Βεβαίως στο Τσερνομπίλ χρειάζονται χρήματα γιατί η σαρκοφάγος αυτή δεν είναι ασφαλή. Επίσης δεν άκουσα ότι θα γίνουν με τα πυρηνικά απόβλητα γύρω-γύρω. Η διάθεση των αποβλήτων αυτών δεν είναι δεδομένη ούτε εξασφαλισμένη. Γι' αυτό Κύριε Ρόιλ, βεβαίω και χρειάζονται έρευνε και μελέτε επιστημονικές, γιατί έχουμε πολύ μικρή εμπειρία με τη μακροχρόνια δράση των ε, ραδιενεργών υλικών. Θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Και τελικά, ξέρετε, η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι η εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας και η συνεργασία με όλες αυτές τις χώρες θα παρακαλούσα για το μέλλον να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να εκμεταλλευτούμε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η επιταγή των καιρών 25 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπεκ σήκωσε γαλάζια κάρτα. Γαλάζια είναι αυτό που σηκώνεται. Μάλιστα, έχετε το λόγο. Καταρχήν πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Λάινε να συμφωνεί. Δέχεστε την ερώτηση. Ωραία. Κύριε Ρούμπεκ, έχετε το λόγο. Το λόγο έχετε μικρόφωνο, δεν έχετε. Ναι. Ευχαριστώ τον κύριο Λάιν. Μίλησε για τα stress τεστ, για τις δοκιμές αντοχής. Θα πρέπει να υπάρχει όμως και συνέχεια. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για αυτό το τομέα που να ασχολείται με αυτό το έργο και να έχει φορτιστεί με τον παροπλισμό επικίνδυνων πυρηνικών εργοστασίων. Σα ευχαριστώ, λέει ο κύριο Λάινε, για την ερώτηση αυτή. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι ο στόχο. Ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των πυρηνικών εργοστασίων. Γιατί εφόσον έχει αυτό επιπτώσει εκτό των εθνικών συνόρων, δεν είναι εθνικό ζήτημα, είναι ευρωπαϊκή η διάσταση και χρειάζεται και ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Και κύριε Επίτροπε, κύριε Τιγκερ, αυτή τη στιγμή δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά θα πρέπει να εργαστεί εργαστείτε προς την κατεύθυνση αυτή να γίνει ανεξάρτητα και αντικειμενικά η Ευρώπη να ε, παρακολουθεί ε, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και ε, να βγάζει και τα απαραίτητα συμπεράσματα όταν χώλει εγκατάσταση γιατί όταν δείξει η δοκιμή ότι δεν είναι ασφαλές το εργοστάσιο είτε να ασφαλίζεται είτε να παροπλίζεται. Ευχαριστώ. Η κυρία Παρβάνοβα από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα της εφαρμογής της ενεργειακής μας στρατηγικής είναι ένα θέμα που απασχολεί τα κράτη-μέλη. Ε, όποια και απόφαση να λάβουμε υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας, το θέμα της ασφάλειας θα πρέπει να μας απασχολεί. Θα πρέπει να έχουμε κοινέ προδιαγραφές ε, για την πυρηνική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί η μόλις η μεραδιενέργεια δεν γνωρίζει σύνορα. Φάνηκε αυτό από το ατύχημα του Τσερνομπίλ και βλέπουμε και τις συνέπειες της Φουκουσίμα. 25 χρόνια μετά τα γεγονότα του Τσερνομπίλ χρειαζόμαστε αποτίμηση των προηγούμενων και των τωρινών κινδύνων ε, για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι μέτρο προστατευτισμού, αλλά μακροπρόθεσμη στρατηγική. Το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων επίση είναι σημαντικό. Τι έχει μείνει από το Τσερνομπίλ, το θέμα των αποβλήτων είναι τρομερό, αλλά και σοβαρό θέμα περιβάλλοντο και ανθρώπινη υγεία. Έχουμε τεράστια πρόκληση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη ασφάλεια για την ε, επεξεργασία ή αποθήκευση των ε, πυρηνικών αποβλήτων. Χρειαζόμαστε μια σαφή και απερίφραστη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Παραβάνοβα. Το λόγο ο κύριος Σιμάνσκι εκ μέρους των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Σας ευχαριστώ. 25 χρόνια μετά την τραγική καταστροφή του Τσερνομπίλ ε, είναι σημαντικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, αλλά μερικές φορές ε, χάνουμε το νόημα. Πριν ε, από 30 χρόνια είχαμε ακόμη και τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικά νομικά μέσα για την εφαρμογή των ε, προδιαγραφών ασφάλειας και είχαμε από τις ψηλότερες ε, παγκοσμίως προδιαγραφές. Βέβαια έγινε μια κατάχρηση για αντιπυρηνική προπαγάνδα στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η πυρηνική ενέργεια μας εξασφαλίζει μια ανεξαρτησία από τις ε, Τρίτε χώρε που είναι προμηθευτές μας. Θα πρέπει να έχουμε και κάποιες θετικές ε, ε, σκέψεις. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές από τις από τα ρωσικά πυρηνικά εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εισάγουμε ηλεκτρικό ρεύμα και αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια δεν τηρούν τις δικές μας υψηλές προδιαγραφές. Έχουμε στο, Καλιγρα... στο Καλίνιγκραντ ή στο... στη Λευκορωσία πυρηνικού σταθμούς που παράγουν ρεύμα που πηγαίνει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε δύναμη και φαντασία πραγματικά για να ε, εφαρμόσουμε τις προδιαγραφές της ασφάλειας και για τις περιοχές αυτές. Η κυρία Χάρμς, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Οτιγκέρ, πιστεύω ότι είναι σωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πάρα πολλά έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του Τσερνομπίλ. Το θέμα είναι κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε αρκετά και κατά πόσον κάνουμε πάντα το σωστό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στον τομέα των συνεπειών στην υγεία εξακολουθούν ε, να υπάρχουν ε, κάποια κενά, πρέπει να καλύψουμε κάποια κενά γιατί υπάρχει αυτή η διαμάχη ως προς ε, τα παραποιημένα στοιχεία που δίνει η Euratom. Αυτή η διένεξη πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το ίμιση της επικράτειά της ε, επηρεάστηκε από το πυρηνικό αυτό ατύχημα οδηγεί στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαφερθεί ιδιαίτερα για το θέμα. Αυτό βεβαίω και είναι αλήθεια. Οι συνέπειες σε διεθνές επίπεδο, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην επικράτεια της πρώην Σοβιετική Ένωσης ή στη Λευκορασία, την Ουκρανία, στη Ρωσία. Πάνω από το ίμιση των ε, συνεπειών προέκυψαν και έπληξαν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο γιατί ακολούθησε όπως γνωρίζετε και η πυρκαγιά και όλες οι άλλες συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν ε, παρακαλώ να αντιμετωπιστείτε τις ε, επιπτώσεις στην υγεία ένα αίτημα που εκφράζεται ιδιαίτερα και πολλοί εργαζόμενοι στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα χαιρούσαν ιδιαίτερα αν η δουλειά του αντιμετωπισόταν διαφορετικά. Τώρα γίνεται παντού λόγος για το νέο μεγάλο περίβλημα, το κάλυμα αυτό. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει καμία ανάλυση κινδύνου για τη σαρκοφάγο υπαριθμών 1. Γιατί το πρόβλημα που υπάρχει επί τόπου δεν το αντιμετωπίζουμε. Πώς είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα να εφαρμόζεται χωρίς να υπάρχει διαφανής ανάλυση κινδύνου. Και πώς μπορούμε παράλληλα να σιωπούμε και μέχρι σήμερα να μην έχει καταστεί δυνατόν ε, τα, ε, καυσίμων να αποφορτιστούν, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τρίτον, από την εποχή του Τσερνομπίλ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν από την Φουκοσίμα βρεθήκαμε πολύ κοντά στο να λιώσει η καρδιά του αντιδραστήρα στο Προυν Σπίτλ, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, εκεί έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η προσωμείωση ακραίων καταστάσεων που έχει, έχει προταθεί τώρα, αυτέ οι προσωμιώσει δεν ενδείκνυνται για να αναλυθεί ο κίνδυνο ο οποίο υπάρχει στου ευρωπαϊκού πυρηνικού αντιδραστήρε. Γι' αυτό λοιπόν σα παρακαλώ θερμά κύριε Έτιγκερ να μας πείτε την αλήθεια. Εσείς υποσχεθήκατε ότι θα υπάρχουν σκληρές τέτοιου είδους προσωμιώσεις, αλλά αυτά τα οποία έχετε καταθέσει μέχρι τώρα δεν είναι σοβαρά. Μετά την καταστροφή του Τσερνομπίλ οι έρευνες της εταιρεία για την προστασία από την ακτινοβολία κατέληξαν στο ότι 1,4 εκατομμύρια άτομα πέθαναν από τις συνέπειες αυτού του πυρηνικού ατυχήματος. Στη Γερμανία φοβόμαστε την ακτοβολία ε, στα παιδιά μας ε, λόγω των ε, βροχοπτώσεων και των μολυσμένων τροφίμων. Η ε, καταστροφή στο Τσέρνομπιλ και στη Φουκουσίμα πρέπει να μας οδηγήσει στο να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα. Ο φόβος ε, ότι οι ανακοινωθήσεις ε, προσωμιώσεις ακραίων καταστάσεων απλά θα αποτελούν άλλοτι για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι πυρηνικές διαδικασίες. Δυστυχώς οι φόβοι αυτοί επαληθεύτηκαν. Άλλε πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν θα ελεγχθούν καθόλου. Κατά πόσον πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, ή για ε, πτώση αεροπλάνου. Οτιδήποτε θα μπορούσε να κοστίσει στις ε, εταιρείε που λειτουργούν στους ποινικού δεν θα εξεταστεί παρότι είναι καθοριστική σημασία για τους πολίτες. Εμείς λοιπόν ζητούμε να υπάρχουν εκτεταμένες ε, τέτοιου είδους προσωμιώσεις από ανεξάρτητους επιστήμονες και αυτό μπορεί να είναι μόνο το πρώτο βήμα, πανευρωπαϊκό βήμα έτσι ώστε να εγκαταληφθεί η πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, η έκρηξη του Τσερνομπίλ ήταν μια καταστροφή, ένα όλεθρο. Αλλά α μην χάνουμε και το θέμα τη της 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από το Τσερνομπίλ σε 23 χρόνια. Και είχαμε και 6.000 ε, περιπτώσει κρούσματα καρκίνου του θηροειδού. Είναι πραγματικά ε, τραγικά αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν είναι τίποτα σε σχέση με το, το φόρο ζωής από τα τροχιά ατυχήματα. Μερικές φορές χρησιμοποιούν μερικοί ως άλλα το Τσερνομπίλ για να ζητήσουν να σταματήσουμε ε, την πυρηνική ενέργεια. Μερικές φορές ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος από αγαθές προθέσεις. Μην ξεχνάμε τι, γίνεται με, τι έγινε με τα βιοκαύσιμα και πώς οδήγησαν σε αύξηση των τιμών των τροφίμων, κάτι που έπληξε τις τρίτες χώρες. Πολύ, πολλά παιδιά λιμοκτονούν στον τρίτο κόσμο, επειδή εμείς, ε, ο δυτικός κόσμος, είχε καθές προθέσεις. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η επίπτωση των ε, αποφάσεων μας στον πραγματικό κόσμο. Γιατί η κατάληψη της πυρηνικής ενέργειας θα είναι ακόμη χειρότερη. Δεν θα έχουμε περισσότερες ανεμογεννήτριες, αλλά η εναλλακτική λύση σε σχέση με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες δυστυχώς θα είναι μαζική λιμοκτονία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορκουνάιτε Μικουλιέν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταστροφή του Τσερνομπίλ μεταξύ άλλων οφειλόταν σε κάποια λάθη στο σχέδιο και κάποιες προβληματικές δοκιμές αντοχής ακραίες συνθήκες που έγιναν. Η πρόσφατη τραγωδία της Φουκουσίμα μας οδήγησε στο να εφαρμόσουμε δοκιμές αντοχής στους πυρηνικούς μας αντιδραστήρες και ευελπιστώ ότι τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών αντοχής θα είναι ικανοποιητικά. Και θα γιατί μην ξεχνάτε ότι η βλάβη στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από ένα πυρηνικό ατύχημα δεν γνωρίζει σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν 25 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ να γίνουν δοκιμές αντοχής σε ακραίες ε, συνθήκες, όχι μόνο στους ευρωπαϊκούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, γιατί βλέπουμε ε, ότι θα κατασκευαστούν νέοι πυρηνικοί αντιδραστήρες στα Λίνιγκρατ, χωρίς όμως να συνοδεύονται ούτε από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε από δοκιμές αντοχής σε ακραίες συνθήκες. Ούτε υπάρχει σαφήνεια ως προς τον τρόπο που σε περίπτωση ατυχήματος και μάλιστα στο Καλίνιγκραντ ο πυρηνικό αντιδραστήρα θα κατασκευαστεί σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε αλληλεγγύη μεταξύ μα και να απαιτήσουμε αντίστοιχε δοκιμέ αντοχή να γίνονται όχι μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στι γειτονικέ χώρε. Και με τη βοήθεια των διεθνών οργανισμών και της γραμματείας του ΣΠΟ θα πρέπει να πετήσουμε σαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις ποιες περιοχές θα επιλεγούν ε, για την κατασκευή τέτοιων εργοστασίων. Ο κύριος Βαλτσίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επίτροποι, η ζήτηση αυτή είναι σημαντική, αλλά έπρεπε να την είχαμε κάνει εδώ και καιρό έχει μεγάλες επιπτώσεις όχι μόνο στο λαό της Ουκρανίας αλλά και στις γειτονικέ χώρες η καταστροφή του Τσενομπίλ και θα γίνουν αισθητά αυτά και από μελλοντικέ γενναίες και δυστυχώς η καταστροφή στη Φουκουσίμα έδειξε ότι μέσα στα 25 αυτά χρόνια ο κόσμος δεν έκανε προσπάθειες ε, για να ε, εκτιμά σωστά και αντικειμενικά τον κίνδυνο από τα πυρηνικά. Ακούμε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι καλύτερη, καθαρότερη και ασφαλέστερη, αλλά οι επιπτώσεις της είναι ε, χειρότερες. Τι θα γίνει και με επιπτώσεις στο μέλλον στις επόμενες γενναίες ανυπολόγιστες. Θα πρέπει κατά βάση και εκβάθρον να αναθεωρήσουμε το πυρηνικό θέμα. Καλωσορίζω τη στρατηγική αυτή για τους ελέγχους και τις προσωμιώσεις των καταστάσεων, αλλά θα πρέπει να είναι συστηματική και όχι τυχαία αυτή η έλεγχη. Θα πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία μας το εξής. Δεν υπάρχει κανένας τομέας που να ρυθμίζεται με σωστό τρόπο, με αυτορύθμιση, αυτοπαρακολούθηση και αυτό δεν ξέρω τι. Θα πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, μια συλλογική αντιμετώπιση και στρατηγική και για τα πυρηνικά και για τις τρίτες ε, χώρες και να παρακολουθούμε για τα εξωτερικά μας σύνορα για να ξέρουμε και τι θα κάνουμε σε περίπτωση που δεν περάσουμε τις δοκιμές ε, τα εργοστάσια. Κυρία Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος που ζούσε γύρω από το Τσενομπίλ και εκείνοι που εργάστηκαν ε, μετά την καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο έπαθαν ε, χρωμελές ζημιές για την υγεία τους και αυτές εξακολουθούν 25 χρόνια μετά και όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και Στη Σουηδία ε, εξετάζουν τα ζώα πριν τα σπάξουν και δοθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, για την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια είναι επικίνδυνη και γι' αυτό χρειάζεται έλεγχος και παρακολούθηση και αξιολόγηση για τους αντιδραστήρες. Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά συστηματικά, ουσιαστικά και σωστά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Και θα πρέπει να αναγκαστεί και η Γαλλία να ακολουθήσει αυτό το δρόμο γιατί δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται. Και πέρα από τις γεωγραφικές ε, σκέψεις θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε και διαφορετική κουλτούρα και διαφορετική νοοτροπία και αντίληψη για την ασφάλεια. Ευχαριστώ κύριο Ζιόμπρο παρακαλώ. Ευχαριστώ. 25 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα του, Τσερνομπίλ αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ποιες είναι οι τραγικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και ζωή αλλά και για το περιβάλλον μια τέτοια πυρηνική καταστροφή. Και είδαμε και πρόσφατα το πυρηνικό ατύχημα και στη Φοκουσίμα. Σίγουρα η ελαττωματική κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα συνέβαλε στο πυρηνικό ατύχημα. Και εμείς προσπαθούμε να ελέγξουμε τους δικείς μας ε, αντιδραστήρες, αλλά το θέμα είναι πώς θα ελεγχθούν και θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια και στους ε, σοβιετικούς αντιδραστήρες. Έχουμε 130 στη Ρωσία και 190 στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες δοκιμές αντοχής, είπαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι δοκιμές αυτές αντοχής δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά και δεν υπάρχουν και κυρώσεις. Ποιες θα είναι οι οι κυρώσει ε, σε περίπτωση αρνητική έκβαση μια ε, δοκιμή αντοχής, γιατί θέλουμε υψηλέ προδιαγραφέ των πυρηνικών ε, αντιδραστήρων, ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί η πυρηνική ενέργεια είναι σημαντική πηγή ενέργεια. Θα πρέπει όμω ταυτόχρονα να αναπτύξουμε και άλλε πηγέ ενέργεια, φυσικό αέριο ή ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, γιατί δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην πυρηνική ε, ενέργεια και να τη θεωρούμε ως κάτι ε, απαραίτητο, απόδραστο. Ο κύριος Σοντή, θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του συναδέλφου και φίλου Μποκούσου Αυσόνικ που ανέλαβε την πρωτοβουλία και υπέβαλε την προφορική ερώτηση για την πυρηνική ασφάλεια 25 χρόνια μετά την καταστροφή του Τζενομπίλ, που ήταν η πιο σοβαρή πυρηνική καταστροφή στην ιστορία τη πυρηνική ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από αυτή την πυρηνική καταστροφή και σα προτείνω τέσσερα συμπεράσματα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε τι καλύτερε προδιαγραφέ ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επηρεάσουμε και του εταίρου μα στα πλαίσια τη παγκόσμια διακυβέρνηση ε, να εξασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες τις καλύτερες προδιαγραφές ασφάλειας χρησιμοποιώντας ε, τις τελευταίες μεθόδους και τεχνολογίες. Επίσης θα πρέπει να πάψει η εμπορευματοποίηση των low cost πυρηνικών αντιδραστήρων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη αλλά και οι, ε, όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να εξασφαλίσουν απόλυτη διαφάνεια των πυρηνικών δραστηριοτήτων. Γιατί θα πρέπει να μπορούν οι πολίτες να, να έχουν αντίληψη του κινδύνου και επίσης θα πρέπει να επιβάλλονται σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση παρατυπιών. Ε, βέβαια, το κόστος της ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος της ενέργειας. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε λοιπόν για να γίνει υποχρεωτικό το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων στις εταιρείες αυτές. Θα πρέπει να προωθήσουμε και τα ερευνητικά μας προγράμματα και την κατάρτιση των επιστημόνων και χαίρομαι για την παράταση του 7ου Ερευνητικού Πλαισίου για την Ευρατόμ για την επόμενη διετία 2012-2013. Κυρία Σαρμπού είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία, μια χώρα που παράγει πυρηνική ενέργεια και όπου ο κόσμος αγωνιά και προβληματίζεται και δεν έχουν απαντηθεί αγωνίες του ως προς τη μακροπρόθεσμη και τις συνέπειες ε, του Τσένομπιλ. Είναι σημαντικό αυτό μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε κυρίως ε, με ε, τη μέτρηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Επιστήμονες πρέπει να κάνουν μελέτες και το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ερευνήσουν όλες τις βλάβες και τις συνέπειες που προκάλεσε στην ανθρώπινη υγεία. Κανονικά θα πρέπει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να κάνει αυτή τη μελέτη. Ωστόσο, υπάρχει σύγκρουση αυτή τη στιγμή μεταξύ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της ε, Διεθνούς Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας για το ποιος θα το αναλάβει. Και φαίνεται να επικρατούν τα συμφέροντα ε, της πυρηνικής ενέργειας. Πριν από 50 χρόνια είχαν συνάψει μια συμφωνία οι δύο οργανισμοί αυτοί και ο Οργανισμό Πυρηνική ενέργεια έχει δικαίωμα, λέει, να αρνείται την πρόσβαση σε στοιχεία στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, γιατί τα θεωρεί απόρριτα. Ακόμα και αυτά είναι σημαντικά για να καταλάβουμε τι επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία. Με άλλα λόγια, ένα οργανισμό που ασχολείται με την προώθηση τη πυρηνική τεχνολογία, αρνείται την πρόσβαση ε, ε, σε δεδομένα για την υγεία αυτή στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ. Πριν από δύο ε, εβδομάδε. πέρασαν 25 ε, χρόνια, ένα τέταρτο αιώνα δηλαδή, από την τραγωδία του Τζερνομπίλ. Θυμάμαι το κομμουνιστικό καθεστώ στη χώρα μου, ε, έδωσε μερικά στοιχεία για την καταστροφή και την 1η Μαΐου είχαμε τις διαδηλώσεις των ανυποψίας των εργατών που δεν γνώριζαν ότι το πυρηνικό σύννεφο περνούσε τότε από την Πολωνία. Έχουμε ε, το θέμα της ε, πυρηνικής ασφάλειας που μερικές φορές ε, εξαιτία έλλειψης πόρων δεν εξασφαλίζεται. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε όμως από την πυρηνική ενέργεια γιατί είναι μοναδικός τρόπος για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ενεργειακού μας ανεφοδιασμού η πυρηνική ενέργεια. Κύριε Κούρσκι, παρακαλώ, μιλάτε ε, ως Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την ατομική ενέργεια, γιατί είναι το καλύτερο, το, ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ενεργειακού μας ανεφοδιασμού. Έχουμε σχέδια για πυρηνικού συντηρητήρε στην Πολωνία, στη Λιθουανία, στη Σλοβακία. Είμαι υπέρ των δοκιμών αντοχή ακραίε συνθήκε. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικέ αυτέ οι δοκιμέ αντοχή και να έχουν έναν συγκυριακό χαρακτήρα, να γίνονται τακτικά. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τη πυρηνική ενέργεια. Αλλά τέτοιε δοκιμέ αντοχή θα πρέπει να γίνουν και στην επικράτεια τη Ρωσία και στι πρώην Σοβιετικέ Δημοκρατίε και στην Ουκρανία και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Το λόγο ο Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Τσερνομπίλ κατέδειξε, όπως βέβαια και το ατύχημα στη Φουκοσίμα, ότι μπορεί κανείς να θεσπίσει όσους κανόνες επιθυμεί. Όμως ε, ε, ο κίνδυνος, στον κίνδυνο πρέπει να συνυπολογίζεται και το ανθρώπινο λάθος κατόπιν τούτου οφείλουμε να πούμε πού ακριβώς βρίσκονται τα όρια της πυρηνικής ενέργειας και σε αυτούς τους υπολογισμούς ε, να μην ξεχνάμε το ανθρώπινο λάθος. Δυστυχώς τότε δεν υπήρξαν αρκετές πληροφορίες και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σοβιετικό σύστημα. Πολλές ε, ε, πληροφορίες οφείλονται ακριβώς σε αυτό το σοσιαλιστικό σύστημα, στον τρόπο που δεν κοινοποιήθηκαν. Και κατόπιν τούτου το σοβιετικό μοντέλο φέρει μεγάλη ευθύνη. Εξάλλου θα πρέπει, ας μην το ξεχνάμε αυτό, οποτεδήποτε υπάρχει ατύχημα να υπάρχει και απαραίτητη διαφάνεια. Τρίτο που θέλω να πω, ε, πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα και από τη δική μου την εκλογική περιφέρεια βοηθούν προσπαθούν να μειώσουν τον πόνο. Καλούν παιδιά από το Τσερνομπίλ. Ε, και ε, αυτό δείχνει λοιπόν ότι με αυτό το υπόλοιπο κινδύνο που υπάρχει δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι όποια και είναι η τεχνολογία. Κύριε Επίτροπε, εγώ θέλω να σας ενισχύσω σε αυτά τα, τις ε, προτινόμενες προσωμιώσεις ακραίων συνθήκων. Ε, τα κριτήρια δεν θα πρέπει να τα ορίζουν μόνο τα κράτη-μέλη. Οι δοκιμές αυτές αντοχής ε, θα πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να επικρατεί η βεβαιότητα ότι αυτό που λέγεται είναι και πραγματικό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να σας ενθαρρύνω να μην ενδώσετε στις απαιτήσεις των Υπουργών και να μιλήσετε με απόλυτη σαφήνεια, να ορίσετε διαυγή κριτήρια έτσι ώστε να υπάρξει και μία βελτίωση. Πρόεδρος, ε, δυστυχώς από ό,τι βλέπω καθυστερούμε για 1,5 λεπτό. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Κάριντς. Κύριε Επίτροπε. Αν κάποιος ε, ζει σε ένα δρόμο που έχει μεγάλη φασαρία, έχει τη δυνατότητα να μετακομίσει, να αποφύγει την ηχορύπανση, έστω και αν ε, μετακομίσει τρία-τέσσερα στενά πιο κάτω. Όμως, στην περίπτωση του Τσερνομπίλ αλλά και στην περίπτωση του Φουκοσίμα πριν από λίγες εβδομάδες διαπιστώσαμε ότι στην περίπτωση της πυρηνικής ενέργειας δεν έχει κανείς την ευκαιρία να μετακομίσει. Η πυρηνική ασφάλεια δεν είναι ένα θέμα περιορισμένου βεληνικούς, είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι χώρες ε, που έχουν σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες αυτές δεν έχουν τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές όπως έχουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να μετακομίσουμε, να απομακρυνθούμε από τους ε, γειτονές μας. Κατόπιν τούτου Εφόσον δεν υπάρχουν παντού τα ίδια αυτηρά κριτήρια, καλό εσάς ε, κύριε Επίτροπε τι ε, προσωμιώσει ε, αντοχής να τις διεξάγετε όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές γιατί είναι απολύτως απαραίτητο οι προδιαγραφές αυτές να εφαρμόζονται και στους γειτονές μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις όμορες χώρες σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Ο κύριος Μαν για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Τόμας Μαν. υπάρχει ο κίνδυνος ακτινοβολίας και γι' αυτό το λόγο αυτοί που ε, πλήγησαν, που ήταν κοντά, θέλησαν να μην βγαίνουν στους δρόμους για ε, να μην εκτεθούν σε πυρηνική ενέργεια. Πρόσφατα είχαμε το ατύχημα στο Φουκοσίμα και ακόμα και η Ιαπωνία με την υψηλή αυτή τεχνολογία δεν μπόρεσε να εφαρμόσει προστατευτικά κριτήρια. Η λύση, για να υπάρχει μια βιώσιμη λύση πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές δοκιμές αντοχής ε, που θα εξετάσουν τις ε, καταστροφές, τις θεομηνίες, τις περιπτώσεις ε, τρομοκρατικής επέκτησης, το ανθρώπινο λάθος. Στη δική μου την χώρα τις αποδίδουν το φόβο, το German Angst όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αυτό όμως είναι λάθος. Θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορα σενάρια γιατί όλα πρέπει να εξεταστούν, να εξεταστούν και ενδεχομένως να καταλήξουν σε ένα δικαιοστάσιο χωρίς να επιβάλλεται οποιαδήποτε τεχνολογία. Η δουλειά της Γερμανικής Επιτροπής Διοντολογίας νομίζω ότι είναι υποδειγματική και μπορούν να την μιμηθούν και άλλοι. Όσον αφορά τους ποινικούς αντιδραστήρες, χρειάζεται ειδική προστασία, ε, να εφαρμόσουμε την σχετική οδηγία, να την συνδυάσουμε με τον κανονισμό περιεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με τον τρόπο αυτό οι κανονισμοί θα αφορούν όλους όσοι βρίσκονται κοντά σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και όλους όσοι έρχονται σε επαφή με πυρηνικά ε, καύσιμα. Τελευταία μου λέξη κύριε Πρόεδρε, ε, πουθενά και που δεν θα πρέπει να υπάρχει συμβασμός για θέματα ασφάλειας. Αυτό ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις ε, όμορες χώρες τις οποίες πρέπει να κερδίσουμε στη δική μας την πλευρά για να λάβουμε από κοινό αποφάσεις. μόνο έναν ομιλητή από κάθε ομάδα θα δεχτώ στη διαδικασία του Catch the Eye. Ο κύριος Μικολάσης, κυρία Χέρτσοκ, Τόιρερ, Χάση, Ράμστορ. Πάσκα, ε, Mrs. Βέρτμαν. Πάσκα. Λυπούμε. I'm sorry. It's not on my list. I do Συγγνώμη κύριε Κολάσκα, αλλά δεν σας είδα στο δικό μου κατάλογο. Λυπούμε ειλικρινά. Λάθος, λάθος κατάλογο. Α, λάθος, λάθος. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Κολάρσκα. Εντάξει, εντάξει, έχετε το λόγο. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, δεν λησμονούμε τα θύματα της ε, πυρηνικής τραγωδίας του Τσερνομπίλ, αλλά δεν ξεχνούμε και τα θύματα της τραγωδίας της Φουκουσίμα και δεν λησμονούμε ούτε την ασφάλεια των, προς, των Ευρωπαίων πολιτών. Και γι' αυτό συζητούμε σήμερα. Στην Ευρώπη το τελευταίο καιρό αυξήθηκε η κοινωνική ανησυχία για την πυρηνική ενέργεια. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις και όλες οι έρευνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Πολωνία 10 με 15% μειώθηκε η υποστήριξη στην πυρηνική ενέργεια και στην κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε τα κριτήρια, τα έξι κριτήρια ασφάλειας των δοκιμών αντοχής που θεσπίστηκα στη Βουδαπέστη. Επίσης, δεν θα πρέπει να ενδώσουμε στις πιέσεις των κρατών που εφαρμόζουν πιο ελαστικά κριτήρια. Επιμένουμε και σε περίπτωση κρίσης, αλλά και σε περίπτωση απλού ανθρώπινου λάθους, να μην ενδώσουμε σε βαλωματικές λύσεις, σε ημίμετρα και σε ε, επίκη κριτήρια. Επίσης, οι δοκιμές αντοχής θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές και για τις χώρες που τώρα αρχίζουν να αναπτύσσουν πυρηνικά προγράμματα. Μιλήσαμε για τις γειτονικέ μας χώρες. Ε, υπάρχουν γειτονικέ χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν πυρηνική ενέργεια, που έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξωτερική διάσταση ενέργεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτέ τι χώρε. γιατί πρόκειται για πυρηνική ενέργεια που επηρεάζει και εμά που έρχεται σε εμά, γιατί και από αυτέ τι χώρε αγοράζουμε είτε φυσικό αέριο είτε ηλεκτρικό ρεύμα και η δική του ε, κατάσταση θα πρέπει να περιληφθεί στην πολιτική μα και να γίνει ένα είδο εξευρωπαϊσμού τη ενεργειακή πολιτική. Σα ευχαριστώ και σα ζητώ και πάλι συγγνώμη που δεν σας είδα προηγουμένως. Στο ΚΑΤΣΤΙΑΙ λοιπόν, ο κύριος Μικολάσιτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά το ατύχημα στο Τζερνομπίλ, αυτή τη φοβερή καταστροφή πριν από 25 χρόνια. 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μέχρι ε, σήμερα υποφέρουν πολύ από τη συνέχεια και τις συνέπειες της ραδιενέργειας που τους ε, προκάλεσαν διάφορες αρρώστιες καρκίνο συχνά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Κοινοβούλιο ασχολείται σήμερα με το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας. Είναι πραγματικά κομβική σημασία. Επίση, κομβική σημασία είναι ότι δυστυχώ χωρί πυρηνική ενέργεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ούτε εμεί στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Κίνα, ούτε στην Ινδία. Όπου έχουν νέα σχέδια κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων, όπω σίγουρα γνωρίζετε. Και στην Ευρώπη θα ήταν υπερβολικό να εγκαταλείψουμε πλήρω κάθε ιδέα κατασκευής νέου πυρηνικού εργοστασίου. Βεβαίω θα πρέπει να παραμείνει κομβική η πυρηνική ασφάλεια κεντρική και να γίνονται αυτές οι δοκιμές αντοχής αλλά και στις γειτονικές μας χώρες και στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία έτσι ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Λέει η Χέτσοκ 25 χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ χρειάζεται να επιδιορθωθεί η σαρκοφάγος και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν οι οικονομικοί πόροι που είναι απαραίτητοι και πόσο δύσκολο είναι να έρθουν από τις ευρωπαϊκές χώρες, ε, τις γειτονικές που ανησυχούν πάρα πολύ ε, για την πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η δέσμευσή μας ε, παραμένει εκεί και μακροπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα παραμένει ο κίνδυνος επιτόπου στο Τσέρνομπιλ και η δημόσια δέσμευσή μας δεν θα πρέπει να είναι μόνο λεκτική αλλά και ε, στην πράξη οικονομική όσο δεν έχει λυθεί το πρόβλημα στο Τσέρνομπιλ. θα πρέπει να βοηθήσουμε και οικονομικά. Αν δεν το καταλάβουμε, θα μείνουμε στα λόγια και σε τίποτα άλλο. Ένα λεπτό παρακαλώ, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τόιρερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Τσένομπιλ μας απασχολεί ακόμα σήμερα 25 χρόνια μετά. Όπως και η Φουκοσίμα θα εξακολουθεί να μας απασχολεί στο μέλλον. Και η αντιμετώπιση με αυτά τα μεγάλα πυρηνικά ατυχήματα δείχνει ότι η πυρηνική ενέργεια συνδέεται με πολύ μεγάλους κινδύνους που ενδεχομένως να μην μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Εδώ χρειάζεται αλλαγή στην οτροπία για την ε, πολιτική, για την ατομική ενέργεια και ε, είναι λανθασμένος ο δρόμος των εθνικών σχεδίων. Θα πρέπει η στρατηγική να είναι διεθνής, να είναι πανευρωπαϊκή. Γι' αυτό υποστηρίζω τον Επίτροπο Ενέργειας που έχει κάνει σημαντικές ε, προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, παρακαλώ όλοι να συμφωνήσουμε στην κοινή αρχή ότι ε, Σημερινέ πυρηνικέ εγκαταστάσεις να είναι ασφαλείς, να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότησή του σε περίπτωση ε, σεισμών, λοιμών, καταποντισμών και λοιπόν θεομηνιών και να είμαστε πάντα υπεύθυνοι. Ευχαριστώ κυρία Χάση για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, 25 χρόνια μετά το Τσενομπίλ δεν έχουμε καθόλου αποτελέσματα ερευνητικά τεκμηριωμένα για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Λαμβάνονται κάποια μέτρα αποσπασματικά και όχι ε, συγχρονισμένα. Ε, προσπαθούν να να μελετήσουν τα περιστατικά καρκίνου του θηροειδού στη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί και να πει ότι Χρειάζεται ευρύτατη μελέτη, επιστημονική έρευνα για την ανθρώπινη υγεία. Ακούμε ότι το Τσερνομπίλ οδήγησε σε λίγα θύματα μόνο, μερικές δουζίνες μόνο. Άλλοι λένε ότι ε, μπορεί να είναι και πάνω από εκατομμύριο ε, τα θύματα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι εικασίες, γιατί δεν έχουμε σαφή επιστημονικά δεδομένα και αποτελέσματα ερευνών. Με τέτοιου είδους μέτρα και με τέτοιου είδους μελέτες θα μαθαίναμε και ποιες είναι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. ομιλητής, κύριος Ράνστορφ. 25 χρόνια, μια επέτειο σλιβερή της θεομηνίας του Τσέρνομπιλ, της καταστροφής, θα πρέπει να θυμηθούμε δύο κράτη που δεν είναι τόσο προσφυλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι η Λευκορωσία και η Ουκρανία. Τα δύο κράτη αυτά σεμνά και χωρίς μεγάλες δηλώσεις και τυμπανοκρουσίες χρηματοδοτούν ε, την επιδιόρθωση ε, του Τσέρνοπιλ χωρίς μεγάλη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Κούβα διότι η Κούβα εδέχθη μεγάλο αριθμό προσφύγων, ιδιαίτερα παιδιά, πάρα πολλά από τις προσβεβλημένες περιοχές και από τις οικογένειες που επλήγησαν από την καταστροφή αυτή. Τους παρήχαν ε, φροντίδα υγείας, περίθαλψη και γενικότερα βοήθεια τότε που ήταν επίσης σε πολύ κακή κατάσταση οικονομικά η Κούβα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κύριε Επίτροπε, οι επιπτώσεις του Τσερνομπίλ, οι είναι γνωστές σε όλους. Λέει κυρία Βέρτμαν. Ε, εκτός όμως από τις ερωτήσεις, περιμένουν και κάποια διδάγματα οι πολίτες. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξηγήσει στον πληθυσμό και τα θέματα της υγείας και τα θέματα τα οικονομικά. Τα γνωρίζει και μετά το Τσερνομπίλ και μετά τη Φουκοσίμα. Ποια μέτρα θα πάρετε σε περίπτωση νέου τέτοιου ε, δυστυχήματος. Διότι οι κινδυνοί στην Ευρώπη είναι αδιαφυσβήτητοι. Το ΙΖΑ 1 που είναι τύπου Φουκουσίμα ε, και ε, είναι στο διάδρομο προσέγγισης για την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Ο κύριος Κέλλη δεν είχε ζητήσει να μιλήσει, αλλά αφού είπατε ότι ζητήσατε το λόγο στο Catch the σας πιστεύω, αλλά έχετε μισό λεπτό για να μιλήσετε. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω τα εξή δύο. Πρώτον, ευτυχώς δεν έχουμε ξεχάσει τα θύματα του Τσέρνομπιλ στη χώρα μου. Ε, υποστηρίζουμε με ε, ε, οργανώσει στα θύματα αυτά και θα εξακολουθήσουμε και στο μέλλον. Και δεύτερον, δράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ και τον Επίτροπο και το είπε και ο κύριος Ρούμπιχ, θα πρέπει μια ρυθμιστική αρχή ευρωπαϊκή να ε, κάνει τις δοκιμές αντοχής και στο μέλλον να ελέγχει όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταστροφή του Τσερλομπίλ μας έδειξε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα σύστημα ενημέρωσης, κοινοποίηση και πληροφόρησης για αυτά τα δυστυχήματα. Οι Σοβιετικοί μας απέκρυψαν το ατύχημα και αυτό είχε σημαντικότατες επιπτώσεις και αρνητικές για τα γειτονικά κράτη. Και στο μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει ε, αυτό το θέμα γιατί είδαμε ότι και στη Φουκουσίμα Βελτιώθηκε μεν ε, η πληροφόρηση, αλλά και πάλι ε, έκρυψαν πληροφορίες. Σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής θα πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο και οι ειδικοί αλλά και οι κοινοί γνώμοι για να μπορούν να αντιδρούν ε, όσο γίνεται καλύτερα με το σωστό τρόπο. Παράδειγμα. Αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, ε, θα πρέπει να είναι πολύ καλή η πυρηνική ασφάλεια, να βελτιωθεί η πυρηνική ασφάλεια. Herr Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το Τσερνομπίλ, ε, Ευχαριστώ να δεχτώ ότι αυτά που προτείνατε και τα αιτήματά μας ε, εισακούστηκαν ε, κυρίως όσον αφορά το θέμα της έρευνας και θα λάβουμε υπόψη μας αυτά που είπατε στα επόμενα βήματα που θα κάνουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε την πλήρη χρηματοδότηση των απαραίτητων τεχνικών μέτρων στην ε, κοινότητα των κρατών και βεβαίως και με συνδρομή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά λοιπόν ε, θέλω να πω σε ευχαριστώ για μια ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση μια συζήτηση που έθιξε και το τι θα γίνει μετά τη Φουκοσίμα. Μετά από αυτή τη συνεδρίαση ε, προβλέπεται επόμενη συνεδρίαση με τους συντονιστές των αρμόδιων κοινοβουλευτικών ομάδων και θέλω να πω το εξή για το Τσέρνομπιλ. Καταρχήν, όσον αφορά αυτέ τι προσωμιώσει αντοχή, εδώ πρόκειται για τέρα εγκόγνητα. Για του πυρηνικού αντιδραστήρε μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχε λάβει χώρα τέτοιου είδου ε, έρευνα, τέτοιου είδου δοκιμέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη σημασία. Θα επηρεάσει το μέλλον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν δούμε λιγάκι τη συνθήκη της Λιζαβόνας που τη συνυπογράψατε και εσείς οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η απόφαση για το ενεργειακό μείγμα ήταν και θα είναι απόφαση των κρατών μελών, δηλαδή των πατρίδων σας, ε, των χωρών από τις οποίες προέρχεστε. Κατόπιν τούτου η απόφαση για τον άνθρακα, ε, για το αέριο, για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας, αυτές οι αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό εμπίπτουν ε, στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για πρώτη φορά προβλέπεται μια ευρωπαϊκή διαδικασία σε θέμα το οποίο κατά τα άλλα είναι αρμοδιότητα κρατών μελών. Προφανώ και αναφέρομαι στο ενεργειακό μείγμα. Έχουμε 14 κράτη-μέλη με πυρηνική ενέργεια και 13 χωρί πυρηνική ενέργεια. Στην Πολωνία, παραδείγματο χάρη μια άκρος ευρωπαϊκή χώρα εκεί ελήφθη η απόφαση ή μάλλον πρόκειται πολύ σύντομα να ληφθεί η μαλλον προκειται πολυ συντομα να η αποφαση για ε, κατασκευή δύο ποινικών αντιδραστήρων. Στην Ιταλία όμως συνέβη το αντίθετο. Εσείς λοιπόν προτείνατε να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή. Θα πρέπει όμως να μου εκχωρήσετε τις νομικές αρμοδιότητες και τις ε, δυνατότητες πρόσληψης ε, προσωπικού. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή είμαι αναγκασμένος να τηρώ τον νόμο. Ακόμα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή ε, Ελεγκτική Αρχή για τα θέματα της ενέργειας ούτε στη συνθήκη της Λισαβόνας ούτε στο οργανόγραμμα της Κομισιόν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν το γνωρίζετε εξίσου καλά όπως και εγώ. Οι προσωμιώσεις ακραίων συνθήκων είναι πολύ σημαντικές. Γιατί, γιατί είναι εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο πλαίσιο αυτών των προσωμιώσεων τα κριτήρια θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Την Πέμπτη λαμβάνει η χώρα αυτή η κέρια συνεδρίαση ανάμεσα σε Ευρωπαίους, Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν κριτήρια ελέγχου ε, παρότι έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις ε, για προσωμιώσεις, ε, για απογοήτευση, για έλλειψη δοκιμών αντοχής. Μα δεν υπάρχουν ακόμα αυτές οι δοκιμές. Την Πέμπτη θα καθορίσουμε τα κριτήρια των δοκιμών. Αυτό που υπάρχει είναι απλά η πρόταση μιας ένωσης, ενός συλλόγου, στον οποίο δεν ανήκει η Κομισιόν. Αναφέρομαι στην Ένωση των Δυτικοευρωπαϊκών αρχών ευρωπαϊκής ενέργειας που συναντήθηκε η ε, συνέλευση αυτή ε, τον Απρίλη. Το τι θα γίνει αυτό βέβαια είναι δικό μας καθήκον. Εδώ θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο χωρίς καμία ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας απόφασης που ήδη ελήφθη αναφέρεται ότι στους ελέγχους δεν συμπεριλαμβάνεται και ο υπολογισμός του ανθρώπινου λάθους. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό, δεν με ικανοποιεί. Γι' αυτό λοιπόν από αύριο το βράδυ ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθυνθώ και στις 27 εποπτικές αρχές ενέργειας, θα τους πω τη δική μου όψη και θα τους πω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλων των ειδών οι κίνδυνοι ανεξάρτητα από πού προέρχονται. Αναφέρομαι σε φυσικά αίτια όπως ε, είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, ε, ε, οι καύσονες, το ε, ιδιαίτερο, ε, ιδιαίτερο κρύο και να λαμβάνεται υπόψη και ο δόλος. Ύπαρξη ή μη. Να λαμβάνονται υπόψη και τρομοκρατικές ενέργειες, ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, όπως επίσης και πτώσεις αεροσκαφών. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα λοιπόν η συζήτηση που έλαβε χώρα μου έδειξε και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σα. Μου έδειξε ότι υπάρχει αρχή μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενδιαφέρονται όλες οι πολιτικές ομάδες για αυτέ τι δοκιμέ αντοχής και για τα κριτήρια που θα καθοριστούν. Βεβαίως, δεν μπορεί κανεί να τα ξεχωρίσει ε, ακριβώς. Στη Φουκοσίμα ποια είναι τα αίτια, φυσικά ή ανθρώπινο λάθος. Εγώ πιστεύω καταρχήν φυσική καταστροφή, σεισμός και τσουνάμι, όμως όσον αφορά στην αντιμετώπιση του κινδύνου, εκεί εμφανίστηκε το ανθρώπινο λάθος, οι ανθρώπινες αδυναμίες. Γιατί και η αδυναμία, η ανθρώπινη αδυναμία έχει παίξει ρόλο μέχρι τώρα στην Ιαπωνία. Ευχαριστώ μετά την Πέμπτη να σας παρουσιάσω τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζετε ότι χρειάζομαι τη συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βεβαίως και την έχω αυτήν, και χρειάζομαι και τη συγκατάθεση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, που αυτή δεν την έχω, την επιθυμώ. Όμως αυτό σημαίνει ότι κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να μου δώσει τη συγκατάθεσή της για τον έλεγχο των κριτηρίων που θα διέπουν τις προσωμιώσεις ακραίων συνθήκων. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στις Βρυξέλλες υπάρχουν ε, συνάδελφοι ε, με ειδική τεχνογνωσία αυτοί εργάζονται πάνω σε όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία όμως θα πρέπει ε, να εκχωρηθούν αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σας υπόσχομαι ότι θα υπάρχει διαφάνεια. Γιατί το Τσερνομπίλ μας δίδαξε ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Και όσον αφορά τις διαπραγματεύσει Τάρτη Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Εγώ αυτά θα σας τα παρουσιάσω με απόλυτη διαφάνεια και θα σας πω επίσης αν τελικά δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Κομισιόν και την Ινσρεκ. Και τότε ίσως αναγκαστούμε να ε, επιστρέψουμε την εντολή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γιατί προσωμιώσεις ακραίων συνθήκων χωρίς τις σωστές προδιαγραφές εγώ δεν θα τις εγκρίνω. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτραπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Ξεκινούμε ήδη με 40 λεπτή καθυστέρηση. Μην το ξεχνάτε αυτό, συνάδελφοι.